Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η σύσταση και τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη-μέλη να περιορίζουν, να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών. Η συγκίτρια είναι η κυρία Φρεντερίκ Ρης. Της δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε μισή ώρα τουλάχιστον ε,